της διαδικασίας ε, που προβλέπονται και θα δημοσιευτούν στα πρακτικά της συνεδρίασής μας. Επίση ο Πρόεδρος της Διασκέψεως των Προέδρων Επιτροπών με ενημερώνει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση ως προς την ε, κατεξουδότηση πράξη πλευρά τη Επιτροπή Γεωργία. Δεν έχει εκφραστεί από μία ομάδα τουλάχιστον ή 40 τουλάχιστον βουλευτέ ε, αντίρρηση και αν δεν εκφραστεί τέτοια αντίρρηση εντό 24 ερών η σχετική σύσταση θα εγκριθεί. Ιδάλω θα πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία. Έχετε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Και φτάνω στην ημερήσια διάταξη των εργασιών.